Λοιπόν, ε, παρακαλώ καθίστε για να μπορέσουμε να αρχίσουμε. Δεν ξέρω ποιος πήρε το λόγο. Μόλις τώρα ποιος μίλησε. Ποιος από σας μίλησε. Ε, κάποια κυρία που μίλησε ισπανικά. Σας ευχαριστώ πολύ που το επισημάνατε ότι πρέπει να αρχίσουμε. Λοιπόν, ξεκινάει η συνεδρίαση και επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μία ανακοίνωση. Λουίς Μάνουελ Ντίας, Γενικός Γραμματέας της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δρα... Α, όχι, με συγχωρείτε, του πρώην Σοσιαλιστικού Κόμματος της Βενεζουέλας, δολοφονήθηκε χθε σε μια πολιτική συνεδρίαση που έλαβε χώρα στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας στη Βενεζουέλα και αυτή ήταν μια συνεδρίαση που έλαβε χώρα από κοινού με την γυναίκα του ε, έγκλειστου δημάρχου του Κάρακας, Καράκας, Λίλιαν Τίντο. Και νομίζω ότι ο πρόεδρος ε, Σούλτς ε, μου είπε ότι η δική μας αντιπροσωπεία έχει το δικαίωμα να μεταβεί επιτόπου ε, περίπου γύρω από την ημέρα των εκλογών ως ε, επίσημη αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου βεβαίως όχι με την έννοια των, ε, της επίσημης αντιπροσωπείας παρακολούθησης των εκλογών γιατί δεν επιτρέπεται αυτό αλλά εν πάση περιπτώσει με κάποια παρεμφερή μορφή Αυτά λοιπόν είχα να σας ανακοινώσω και περνάμε στο θέμα της Βενεζουέλας. Έχουμε από 4 μέχρι 7 Νοεμβρίου ε, προκαταρκτική αντιπροσωπεία Μάρτο Ρίγκο Μάουρα είναι τα μέλη της αντιπροσωπείας και θα ήθελα να μας ε, ενημερώσετε σύντομα για την αποστολή αυτή. Δεν ξέρω ποιος από εσά τους τρεις θα το κάνει. Παρακαλώ, εσείς. Καλή σας μέρα και ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο Γαμπρίελ Μάτο θα συμπληρώσει αυτά που θα πω εγώ δίχως άλλο, αλλά αρχίζω. Όπως γνωρίζετε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Φεβρουάριο του 2014 ε, να ένα ψήφισμα ε, με το οποίο επιτρεπόταν μια ερευνητική κατά κάποιο τρόπο αποστολή στην Βενεζουέλα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να διαρευνήσει εκεί την κατάσταση. Αποφασίστηκε να πάνε 12 άτομα από διάφορες πολιτικές ομάδες και για μήνες προσπαθούσαμε με τον πρόεδρο Μπροκ επικεφαλής να πετύχουμε άδεια από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας για να υλοποιηθεί η επίσκεψη αυτή, αλλά δεν κατέστη δυνατό. Τελικά αποφασίσαμε να πάμε σε μια πιο μικρή ε, αντιπροσωπεία και όντω τρία μέλη, τρει τρεις ευρωβουλευτές από τρεις κοινοβουλευτικέ ομάδες, ο κύριος Μάτο από το ΕΛΚΟ, ο κύριος Μάουρα από το ΑΛΔΕ και εγώ ο ίδιος από τους σοσιαλιστές πήγαμε τελικά στην Βενεζουέλα. Πριν πάμε εκεί. Προσπαθήσαμε να πετύχουμε άδεια, επίσημη άδεια δηλαδή, από πλευρά τη κυβέρνηση της Βενεζουέλα, η οποία όμως δεν ήταν διατεθειμένη να μας τη δώσει. Ούτε επίσημη θεώρηση για την αποστολή αυτή. Και έτσι τελικά αποφασίσαμε, δεδομένου ότι η προκλητική εκστρατεία άρχιζε και θεωρήσαμε απαραίτητο να φέρουμε σε πέρα στην αποστολή μας, να πάμε. Οπότε, με τον ε, πρόεδρο Μπρόκ αποφασίσαμε έτσι τρεις ευρωβουλευτές να πάνε σε διερευνητική αποστολή στη Βενεζουέλα. Πρέπει να σας πω ότι παρόλο που δεν είχαμε την επίσημη άδεια και δεν ε, μας υποδέχτηκαν ε, κυβερνητικοί, αντίθετα έγιναν κάποιες δηλώσεις και πολύ φιλικές, δεν είχαμε όμως τελικά πρόβλημα να μετακινηθούμε με απόλυτη ελευθερία και με ασφάλεια Όσο καιρό βρισκόμασταν εκεί, μπορέσαμε να έχουμε όλες τις επαφές που θέλαμε να έχουμε και είχαμε προβλέψει να κάνουμε. Τα συμπεράσματα τώρα τα έχετε και στην έκθεση που σας ε, μοιράσαμε. Με δύο λόγια είναι τα εξή. Πρώτον, όλες οι οργανώσεις με τις οποίες ήρθαμε σε επαφή και ήταν πραγματικά πάρα πολλέ από την κοινωνία των πολιτών και τον πολιτικό κόσμο της Βενεζουέλας, οικονομολόγους, πολιτολόγους, ε, αναλυτές πολιτικούς, δηλαδή ακόμα και με τον νούντσιο του Βατικανό, με εσωτερικές επιτροπές παρατήρησης των εκλογών, με κυβερνητικές οργανώσεις, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφους, μέσα ενημέρωσης. Ουσιαστικά ήρθαμε σε επαφή με ολόκληρη την ε, πολιτική ε, κοινωνία και την κοινωνία των πολιτών αλλά όχι με κυβερνητικούς. Εμείς ζητήσαμε να βρεθούμε με το Υπουργείο Εξωτερικών, με την Εθνική Εκλογική Επιτροπή ζητήσαμε να έχουμε συναντήσεις με διάφορες αρχές της κυβέρνησης της Βενεζουέλας αλλά δεν ε, δέχτηκαν να συναντηθούμε μαζί μας. Οπότε η έκθεσή μας δεν περιλαμβάνει και τα συμπεράσματά μας δεν περιλαμβάνουν την άποψη των κυβερνητικών. Οι μαρτυρίες όμως που πήραμε ε, κατέληγαν ομόφωνα σε αυτά που θα σας πω τώρα. Πρώτον, συμπέρασμα. Ο λαός της Βενεζουέλας περνάει μια δύσκολη περίοδο. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για μια χώρα που έχει πολύ υψηλό δίκτυο εγκληματικότητας. 25.000 δολοφονίες στον χρόνο λαμβάνουν χώρα εκεί. Υποφέρει από μια οικονομική κατάσταση επίσης, πολύ δύσκολη, με έναν πληθωρισμό που είναι κοντά στο 200% έχει συναλλαγή με το δολάριο μία επίσημη τιμή και μία ανεπίσημη τιμή που προκαλούν μια κατάσταση που δεν είναι πολύ καλή για τους ε, πολίτες. Καταλαβαίνετε ότι για να αγοράσουν προϊόντα πρώτης ανάγκης δυσκολεύονται. Επίσης τα νοσοκομεία δεν προμηθεύονται τα όσα χρειάζονται. Ο κόσμος δηλαδή υποφέρει. Έπειτα αυτό το οποίο διαπιστώσαμε είναι ότι ο λαός της Βενεζουέλας τουλάχιστον οι οργανώσει με τι οποίε συναντηθήκαμε μα είπαν ότι δεν μπορεί εύκολα να μεταφέρει την απόψή του ο Οπότε η επίσκεψή μα ήταν πολύ καλή, σε μια πολύ καλή στιγμή, γιατί ο κόσμο είχε την ανάγκη να μιλήσει, να περιγράψει αυτά που ζει. Τώρα από πλευρά ε, δημοκρατικών ε, δομών στη Βενεζουέλα θα θυμόσαστε ότι στι προεδρικέ εκλογέ πριν από δύο χρόνια ο κύριο Μαδούρο κέρδισε με μικρή διαφορά. Ε, 223.000 ψήφοι ήταν η διαφορά ανάμεσα στους δύο υποψηφίους, κάτι το οποίο οδήγησε σε διαδηλώσεις που με τη σειρά τους κατέληξαν σε βία στους δρόμους με 43 νεκρούς μεταξύ των διαδηλωτών και των αστυνομικών. Σίγουρα υπήρξε βία, σίγουρα υπήρξε καταστολή από πλευρά της αστυνομίας, δεν θα κρίνουμε εμείς βέβαια τα πράγματα. Το βέβαιο είναι όμως ότι από τη στιγμή αυτή και μετά η κατάσταση επιδεινώθηκε και οδήγησε στο να μην μπορέσουν να αναλάβουν τα καθήκοντά τους διάφοροι εκλεγμένοι ε, βρέθηκαν στη δικαιοσύνη διάφοροι εκλεγμένοι, δήμαρχοι και υπεύθυνοι πολιτικών κομμάτων, οι ηγέτες των φοιτητών που δεν συμφωνούσαν με την κυβέρνηση, σκλίνανε τη στάση της η κυβέρνηση απέναντι στην αντιπολίτευση και η αντιπολίτευση τελικά συγκεντρώθηκε γύρω από αυτό που ονόμασαν Δημοκρατική Ενότητα και αυτή ακριβώς η Δημοκρατική Ενότητα αποτελεί σήμερα την αντιπολίτευση στη Βενεζουάλα. Τα συμπεράσματά μου λοιπόν είναι τα εξής. Οι ανοιχτές ε, δίκες, δικαστικές δίκες δηλαδή, της αντιπολίτευσης δεν είχαν τις εγγυήσει που πρέπει να έχουν σε ένα δημοκρατικό κράτος. Δεύτερον, δεν μπορούμε να πούμε ότι η δικαστική εξουσία είναι εντελώ ανεξάρτητη από την κυβέρνηση στη Βενεζουέλα, δυστυχώς. Τρίτον, η εκλογική διαδικασία που προχωράει εν ώψη των εκλογών της 6ης Δεκεμβρίου επηρεάζεται πώς να το πω, από άνισες συνθήκες όσον αφορά τους υποψηφίους. Δηλαδή αυτοί της κυβέρνησης έχουν πιο εύκολα πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης από τους άλλους κλπ. Οπότε αυτό επηρεάζει την εκλογική διαδικασία. Παρόλο που, πρέπει να το πω και αυτό, η παρατήρησή μας εν ώψη των εκλογών αυτών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει ε, απάτη. Δηλαδή τεχνικά είναι πολύ προηγμένο το εκλογικό σύστημα στη Βενεζουέλα και δεν επιτρέπει παρατυπίες. Και τελειώνω με το εξή Πρόεδρε. Η αντιπολίτευση και η κυβέρνηση βρίσκονται σε αντιπαράθεση αυτή τη στιγμή. Από τις 6 Δεκεμβρίου η Βουλή θα είναι κατά πάσα πιθανότητα αντίθετη με τον Μαντούρο, οπότε η συνύπαρξη θα είναι δύσκολη σε αυτή τη χώρα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν, και αυτή είναι η πρότασή μου, πρέπει να πάει και να συμμετέχει σε αυτή την πολιτική διαδικασία. Είναι πολύ σημαντικό η αποστολή αυτή, η αντιπροσωπεία που αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πάει στην Βενεζουέλα, να πάει τελικά. Και η σύσταση που έγινε τότε για επίσκεψη στη χώρα να ισχύσει πολιτική παρουσία εκεί και όχι ως παρατηρητές των εκλογών. Την επόμενη εβδομάδα πρέπει να γίνει αυτό. Χρειάζεται η πολιτική διαδικασία της Βενεζουέλας στη βοήθειά μας. Αυτά, Πρόεδρε. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε. Εσείς. Ναι, συμφωνώ απόλυτα με τόσα είπε ο συνάδελφος, αλλά θέλω να υπογραμμίσω κάτι. Είπατε ο Λούις Μανουέλ Φεντίας δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια μιας ε, πολιτικής ε, εκδήλωσης. Αυτό δεν είναι απλώς μια ανακοίνωση, είναι η πραγματικότητα που ζει σήμερα η Βενεζουέλα. Πρόκειται για ένα καθεστώς σε μια χώρα που όσες φορές και αν ψηφίσει τελικά καταλήγει να είναι αντιδημοκρατική η κατάσταση και είναι αντιδημοκρατική γιατί δεν υπάρχει ελευθερία. Σήμερα στη Βενεζουέλα είναι προφανές ότι δεν υπάρχουν ελευθερίες ούτε εξουσίας, ούτε τύπου, ούτε για να γίνουν οι εκλογές κάτω από ισότιμους όρους για όλους. Δεν είναι ελεύθερε αυτές οι εκλογές, δεν είναι ελεύθερε για την αντιπολίτευση. Το είδαμε και σήμερα, είναι αποκορύφωμα πράξεων που διαδέχονται μία την άλλη. Είδατε ότι κι άλλους τον δήμαρχο τον υποδέχτηκαν με πυροβολισμούς για παράδειγμα. Τον Πιθάρο. Αυτή είναι η πραγματικότητα λοιπόν σήμερα στη Βενεζουέλα η αντιπολίτευση ή είναι στη φυλακή ή δεν μπορεί να συμμετάσχει στις εκλογές εξαιτία των διαδικασιών. Και όλοι φοβούνται μήπως δολοφονηθούν ή απαχθούν από την αντιπολίτευση. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ από τον Πρόεδρο να κάνει ό,τι μπορεί ώστε να πάμε στις 6 Δεκεμβρίου στη Βενεζουέλα. Μία αντιπροσωπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δηλαδή. Και να μην γίνονται επιλεκτικά προσκλήσεις που το μόνο αποτέλεσμα που έχουν είναι να νομιμοποιούν την ε, κυβέρνηση χωρίς να πρέπει. Συνεπώς, η κατάσταση αυτή στην Βενεζουέλα πρέπει να αλλάξει. Πριν από λίγες μέρες κάποιοι αρνήθηκαν το βραβείο Ζαχάροφ στην αντιπολίτευση της Βενεζουέλας, παρόλο που κάποιοι από αυτούς έχουν δολοφονηθεί στους δρόμους. Ευχαριστώ. Και ήταν πολιτικές δολοφονίες. Ευχαριστώ. να κάνω μια πρόταση. Δεν ε, πρέπει να συζητάμε όλη την ώρα Βενεζουέλα γιατί έχουμε και την ψηφοφορία. Νομίζω λοιπόν ότι όσοι θέλουν τώρα να μιλήσουν να το κάνουν και μετά να συνεχίσουμε τη συζήτηση ε, όταν έχουμε, αν έχουμε τελειώσει πιο ε, σύντομα με την ψηφοφορία. Έτσι λοιπόν ε, θα, θα χρειαστεί να περάσει η ψηφοφορία αργότερα. Όποιος θέλει λοιπόν να λάβει το λόγο θα γράψουμε το όνομά του και θα γίνει συζήτηση μετά την ψηφοφορία. Εντάξει. Πριν από οτιδήποτε άλλο, θέλω να πω ότι οι πληροφορίες που είχαμε ε, είναι αξιόπιστες γιατί ήρθαν από δημοσιογράφους όπως είπε και ο κύριος ε, Μάτο δεν ήταν ακριβώς σε προεκλογική εκστρατεία δεν γίνονται έρευνες όπως θα έπρεπε για να καταλήξουμε σε σωστά συμπεράσματα. Συνεπώς, δυστυχώς έπεσαν οι τόνοι. Οι πληροφορίες που φτάνουν σε μας είναι αντιφατικές. Απ' τη μια λένε οι δημοσιογράφοι ότι μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους από την άλλη όχι. Οι αντιπρόσωποι μας εκεί δεν μπορούν να μιλάνε για ομοφωνία γιατί επισκέφτηκαν και συναντήθηκαν με ορισμένους μόνο, όχι με όλους. Έπειτα όσον αφορά την οικονομία. Λέτε ότι η ένδια μεγαλώνει εκεί. Η φτώχεια επιδεινώνεται. Ε, πράγματι. Αλλά αυτό έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Συγχρόνως όμως υπάρχει ένα κράτος εκεί που προσπαθεί να διορθώσει τα πράγματα. Είπατε για την στήριξη 25% του Μαντούρου. Μα αυτό είναι από δημοσκόπηση. Και είναι απόλυτα φυσιολογικό σε οποιαδήποτε χώρα. Όταν κάποιος με μια τόσο μικρή διαφορά κερδίζει, είναι λογικό να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα τώρα. Λέτε επίσης ότι το εθνικό εκλογικό σύστημα κάνει καλά τη δουλειά του, ότι πάνε καλά εκλογές. Απ' την άλλη όμως λέτε ότι όχι. Υπάρχουν ε, πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά στην προεκλογική διαδικασία. Ε, τελικά ή ε, το ένα ή το άλλο. Μα τι γίνεται. Ή μήπω είναι η Βενεζουέλα η πιο βία χώρα του κόσμου. Όχι, η Ονδούρα είναι σύμφωνα με την τις, ε, τα αποτελέσματα που έχουμε από έρευνε. Έπειτα, για τους δημοσιογράφους, συνεδεθήκατε με κάποιου, αλλά όχι με κάποια οργάνωση. Έπειτα, στην ε, Κολόμβια έχουν δολοφονηθεί περισσότεροι. Μιλάτε για τον τύπο. Μα πάντα. Έτσι δεν λέμε στην Βενεζουέλα. Υπάρχουν εκατόν τόσες τηλεοράσει από τις οποίες 68 σε χέρια ε, ιδιωτών, είναι ιδιωτικά κανάλια. Και μεταξύ αυτών και 18 πιο σημαντικέ. τελεσούρο, κλοβιζιόν κλπ. Το 80% των καναλιών αυτών είναι απόλυτα ανοιχτά στην αντιπολίτευση. Τα στοιχεία που δίνεται δεν είναι σωστά. Θέλω να υπενθυμίσω τι έκανε ο κύριος Λόπες. Υπάρχουν αμαγνητοσκοπήσεις πήγε στην πρεσβεία της Κούβας και παράνομα ε, προχώρησε στην απαγωγή ενός αξιωματούχου. Λοιπόν, πού βασίζεται σε οποιαδήποτε δημοκρατική χώρα ένας πολιτικός ο οποίος επιτίθεται σε μία πρεσβεία που προστατεύεται από τις εμβάσεις της Γέννηση. Απάγει έναν ε, υπουργό, βρίσκεται στη φυλακή, όμως πήρε άφεση το 2008. Αυτός είναι ποματιάς Αφήστε με να μιλήσω κύριε Νάρ. Δεν ενοχλώ κανέναν όταν μιλάει, δεν του κόβω το λόγο. Αφήστε με λοιπόν να ολοκληρώσω. Ευχαριστώ πολύ. Αν έχουμε την ευκαιρία και είμαστε γρήγοροι θα συνεχίσουμε την ε, συζήτηση αργότερα. Σας είπα συνάδελφε ότι κάποιος έχασε τη ζωή του. Ήταν ε, ε, αυτό... Ήταν ένας πολιτικός κρατούμενος, ήταν η χείρα του μαζί, του μαζί και σε μια επίσκεψη που έγινε σκοτώθηκε ο άνθρωπος αυτός. Νομίζω λοιπόν ότι δεν θέλουμε να ε, μπούμε σε αυτή τη θέση και να εκπροσωπούμε τους πιθανούς ε, ε, δολοφόνους σε μια χώρα τώρα που έχει και τόσο μεγάλη εγκληματικότητα, ποσοστό εγκληματικότητας. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα στην ψηφοφορία. Διαδικαστικό, διαδικαστικό πρόεδρε. Δεν έχετε το λόγο. Λέμε ότι τώρα ψηφίζουμε και αν έχουμε χρόνο μετά θα συζητήσουμε. Παρακαλώ, Όχι. Όχι, δεν έχετε το λόγο. Ε, είπαμε θα ψηφίσουμε και μετά. Ξεκινάμε την ψηφοφορία. Και μετά μπορούμε να συζητήσουμε παρακάτω και εγώ θα, συζητήσω, θα συμμετάσχω στη συζήτηση έτσι. Ε, ερχόμαστε τώρα στην ψηφοφορία για την έκθεση της Κίνας. 324 ε, και η τροπολογία 324 Παρακαλώ, σταματήστε εκεί πέρα, κυρίε. Ε, θέλουμε να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Όσοι έχετε κάποια συζήτηση να κάνετε, παρακαλώ να βγείτε έξω. Πρότεινε η ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών να έχουμε μια συμβαστική τροπολογία τη 13 να την ε, επεκτείνουμε με μια πρόταση τροπολογίας η οποία θα αποφύγει να υπάρχουν ε, παρεξηγήσεις στην ΙΤΑ. Ε, θέλει κάποιος να πει κάτι, υπάρχει κάποια αντίρρηση στο να μπει αυτή η νέα ε, τροπολογία. Για να μην συζητάμε και έχουμε προβλήματα, νομίζω ότι καλό είναι να τη βάλουμε. Βλέπω ότι κανείς δεν έχει αντίρρηση, άρα την αποδεχόμαστε και θα την ψηφίσουμε μαζί με την 13. Ξεκινάμε λοιπόν. Θέλει να κάνει κάποια παρατήρηση ο εισηγητής πριν ξεκινήσουμε με την ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Σύντομα. Είμαι εισηγητής. Ήθελα θέλω να πω ότι σε επικοδομητικό κλίμα έγιναν οι συνεννοήσεις και το αποτέλεσμα είναι καλό. Das ist doch schon mal αυτό είναι καλό να το ακούμε. Λοιπόν, πάμε στην συμβαστική τροπολογία 9. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 167 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 177 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 178 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Πάμε στην 179 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Der Antrag 180, wer ist dafür? 180 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 189 υπέρ κατά αποχές ποιος είναι υπέρ 189 εγκρίθηκε η συμβαστική 10 άρα 189. Παονόβα είναι η τροπολογία. Κύριε Γκάλερ, είναι η λίστα ψηφοφοριών του ΕΛΚ. Καλημέρα. Ποιος είναι υπέρ. 189 ψηφίζουμε. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 191 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίνεται. 193 υπέρ. Κατά. Αποχές. Για να κάνουμε ένα τσεκ. Hmm? Ist angenommen mit 29 Εγκρίνεται με 29 ψήφους, ψήφους υπέρ, 25 κατά. Πάμε λοιπόν στην 194 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ψηφίσουμε. Ηλεκτρονικά. Ε, τη της 28 υπέρ, 29 κατά, απορρίπτεται. 195 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 196-197 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 198 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε. πέρα της ψηφοφορίες. 36 υπέρ, 27 κατά εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 που είναι. Που είναι η 12. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13 ε, με την ε, προφορική τροπολογία που σας παρουσίασα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 16. Μόλις την κάναμε. Ωραία. Πάμε στην 203. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 204. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 205. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 206. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 207 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 199 την είχαμε εγκρίνει όχι 209 ε, υπέρ κατά απορρίπτεται 210 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται για... Να ελέγξουμε. Η 11. Υπέρ. Την 10. Όχι, η 10 την εγκρίθηκε. Την 11 τώρα. Την 11. Υπέρ. 211. Κατά. Εγκρίνεται. 212 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε. Τη 212. Πέρας της ψηφοφορίας. 35 υπέρ, 26 κατά εγκρίνεται. 214 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 215 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 216 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε. Ωραία, ας ελέγξουμε την 216. Πέρα της ψηφοφορίες; 32 υπέρ, 37 κατά, απορρίπτεται. Να πω όμως ότι στο ΕΛΚ ε, έχουμε δύο παραπάνω ψήφους. Από τους ε, φιλελεύθερους πάντοτε είστε παραπάνω. Παρακαλώ στο ΕΛΚ να το ρυθμίσετε αυτό, να έχουμε δύο λιγότερους. Πάμε στη 214. Ε, συγγνώμη, στη 217 υπέρ. Κατά αποχές κρίνεται. 219 υπέρ. κατά αποχές απορρίπτει. 220 υπέρ κατά απορρί... εγκρίνεται υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 232 υπέρ και 31 μαζί εγκρίνεται 233 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 18 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 251 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 19 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική 20. Παρακαλώ. Δεν ακούγεται ο μιλητής, είναι εκτός μικροφώνου. Ποιος θέλει να πόσχει. Ωραία, ευχαριστώ. Θα το γράψω στην ιστορία. Συμβαστική 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. 261 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 262 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 74-76 υπέρ ε, αποχές απορρίπτεται 64-65 συγγνώμη 266 ε, υπέρ κατά αποχές το ε, ΕΛΚ και οι σοσιαλιστές είχαν λιγότερους. 266. Επαναλαμβάνω υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 21 αν το βλέπω σωστά. Σωστό. 273 του Γκόμες. Ποιος είναι υπέρ. Δεν είναι τίς γόμες, δεν είναι να κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ελέγχουμε. Πέρας της ψηφοφορίας. 35 υπέρ, 29 κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 21 λοιπόν υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 274 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 278, 79, 280, όλα μαζί είναι παρόμοια σε αυτές οι τροπολογίες, οι ίδιες μάλλον. Γιατί τους ίδιους βέθους, ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ο 285 τώρα. Σωστά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε. Πέρα της ψηφοφορίας. 16 υπέρ, 47 κατά, απορρίπτεται. Πάμε στην 22, συμβαστική 22 υπέρ, κατά, αποχές, συγκρίνεται. 290 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 294 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 295 υπέρ για την 94 να ελέγξουμε πέρα στις ψηφοφορίες Σαράντα υπέρ, 22 κατά, εγκρίνεται. 2,95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνες, 300 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 301 παρακαλώ υπέρ κατά αποχές ε, και εδώ δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα ξανά γιατί 301 υπέρ παρακαλώ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα Έκλεισε η ψηφοφορία. Ε, το αποτέλεσμα 21 υπέρ, 35 κατά, δύο αποχές, απορρίπτεται. Πάμε στη συμβαστική 23. Υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά περνάμε στην 303. Υπέρ παρακαλώ. 303. 303. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται του κυρίου Τόκες 308 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 312 313 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 316 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η συμβιβαστική 25 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 329 παρακαλώ, ε, υπέρ, Η 324 αποσύρθηκε. και αυτή αποσύρθηκε. Έτσι τουλάχιστον αναφέρεται στο δικό μου τον κατάλογο. Οι 322 και οι 323 αποσύρθηκαν, που σημαίνει πάμε στην 329. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 311 υπέρ. Συγγνώμη, λάθος λέει ο πρόεδρος. 331 υπέρ της 331 του κυρίου Μποργέζιο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η συμβαστική 26 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Που σημαίνει πάμε στην 336 υπέρ. Κατά. Ξανά. Υπέρ της 336 παρακαλώ. Κατά Για, να, για δες, περίεργη συμμαχία αυτή. Ούτε, δεν το έχω ξαναδεί ποτέ αυτό. Αυτή τη συμμαχία που δημιουργήθηκε για να ψηφιστεί και είναι η στιγμή αξέχαστη. Κάπως πρέπει να συγκρατήσουμε αυτή τη μοναδική συμμαχία. Από άκρα δεξιά μέχρι τον κύριο Λάινεν έφτασε αυτή η συμμαχία. Τέλος πάντων, έκλεισε λοιπόν η ψηφοφορία. Η 36 με 26 το αποτέλεσμα εγκρίνεται. 3.37 υπέρ, κατά, αποχές απορρίφθηκε. Συμβαστική 27 παρακαλώ, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 3.44 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η 3.45 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται η 327 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 347 <laughs> ψηφίζουμε για την 347 υπέρ κατά αποχές ε, ε, σας το είπα ότι θα απορρίπτεται μου ξέφυγε και το είπα το προέταξα κατά κάποιον τρόπο. Πάμε στην επόμενη. 366 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 348 υπέρ κατά γιατί 348 ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. η 348 του κυρίου Μπίτικοφερ. Αυτήν ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Μισό λεπτό παρακαλώ. Ξανά. Γιατί σταματήσαμε την ψηφοφορία πολύ νωρίς, άρα επαναλαμβάνουμε. Παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Αποτέλεσμα 25-35. Απορρίφθηκε η τροπολογία. Άρα ε, ο κύριος Λάινεν ε, κτά και άλλες ευκαιρίες ενισχύει τη θέση του 349 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται εγκρίθηκε η 349 Οι άνθρωποι εδώ, λέει ο πρόεδρο εκ των δεξιών δεν καταλαβαίνουν το μεγαλείο του. Λέει ο πρόεδρο έκλεισε η ψηφοφορία. Λοιπόν, 35 υπέρ, 22 κατά, 4 αποχές, εγκρίνεται. Τώρα, Σαφχάουζερ, 350 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 351-352 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 353 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήτευση παρακαλώ Έκλειση ψηφοφορία 33 υπέρ, 31 κατά, 3 αποχές, εγκρίνεται. Πάμε στην 354 ε, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 355 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η συμβαστική 28 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 358 υπέρ κατά 358. Ξανά, ποιος είναι υπέρ της 358 παρακαλώ. Υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 360 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 364 υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση. Νομίζω όμως ότι εγκρίθηκε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Αποτέλεσμα 36 υπέρ, 29 κατά ή 365 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 366 υπέρ κατά αποχές γκρίνεται, η 367 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 368 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 369 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 370 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 371 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 372 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ Έκλεισε η ψηφοφορία και η τροπολογία εγκρίθηκε. Πάμε τώρα στην 373, 374, 375, 376 και 377 σε αυτές τις τροπολογίες παρακαλώ που είναι όλες ταυτόσιμες που από ό,τι φαίνεται είχαν όλοι ταυτόχρονα την ίδια επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος για να είναι όλες ταυτόσιμες τροπολογίες. Ποιος είναι παρακαλώ υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση. Λοιπόν, η ψηφοφορία απορρίφθηκε. Άρα δηλαδή οι προσευχές όσο ε, θερμές και να ήταν δεν απέδωσαν, λέει ο πρόεδρος. Πάμε στην 378 υπέρ παρακαλώ. Ε, με σχόλια 387 υπέρ κατά. Ό, όχι 378, ναι 378 με σχόλια υπέρ κατά Ηλεκτρονική επανήθελψη για την 378 έκλεισε ψηφοφορία. 12 με 50 το αποτέλεσμα. 379 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Οι επόμενες 380, 381, 382, 383. Κοιτάξτε, καλύτερα στην αλφή να τα βρουν εκ των προτέρων για να μην φαίνεται ότι έχουν όλοι το ίδιο συντάκτη, λέει ο πρόεδρο. Ποιο είναι υπέρ αυτών των τεσσάρων τροπολογιών κατά αποχέ ηλεκτρονική επαλήθευση, παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Πάμε τώρα στην επόμενη, στην 387, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 388, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 389 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 3 3.97 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Πάμε τώρα στην 399 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 403 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Εγκρίνεται λοιπόν η τροπολογία αυτή. Λοιπόν, λέει ο Πρόεδρος, δυστυχώς ε, κάναμε ένα λάθος. Δεν ψηφίσαμε για την 384 και την 385. Πάμε πίσω λοιπόν. Ποιος είναι παρακαλώ υπέρ της 384. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η 385 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. Έκλεισε η ψηφοφορία. Λοιπόν, 404 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 407 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 408 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 409 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 4.12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4.13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4.14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4.15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 16 4.16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4.19 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 4.20 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 4.22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 423 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 424 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 425 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 421 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε πέρας της ψηφοφορίας 26 υπέρ 39 κατά απορρίπτεται 417 ε, υπέρ κατά ελέγχουμε Εγκρίθηκε η 421, οπότε καταπίπτει η 417. 418 λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε. Πάλι η ίδια εικόνα σε όλη την αίθουσα. Πέρα τη ψηφοφορία. Πάλι το ΕΛΚΑ έχει έναν παραπάνω. Πάλι ένας παραπάνω. Ο Μπλένκοβιτς. Ξεκάθαρα. Πέρα της ψηφοφορίας. 33 υπέρ, 31 κατά, ε, εγκρίνεται και δύο εποχές. 426 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 427 υπέρ, κατά, αποχές, ελέγχουμε. Πέρα της ψηφοφορίας 42 υπέρ, 23 κατά. Εγκρίνεται. 428 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 34 34 υπέρ. Πού είναι. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Είναι στο κάτω μέρος της σελίδας 14. Πάμε στην 435, σωστά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 36 ε, υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε την 436 Αμπετίνη, ποιος είναι, ηλεκτρονικά ψηφίζουμε σχεδόν κλείνει η ψηφοφορία ναι έκλεισε απορρίπτεται 440. 440. Συγγνώμη, 438 πρώτα. Εγκρίνεται. Με την συμβαστική οπότε, το 438 απορρίπτεται ομόφωνα 438 κατά αποχές απορρίπτεται. 440 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 441 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 442 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 449 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 453 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 454 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. 40 υπέρ, 24 κατά. εγκρίνεται. 459 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε. Πέρας της ψηφοφορίας. Με 27 ψήφους υπέρ και 26 κατά και 12 αποχές εγκρίνεται η 460 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 463 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 465 και 66 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε. Πέρας της ψηφοφορίας. 35 υπέρ, 22 κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική 31 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 472 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 32 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 479 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 481 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 484 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ. Συμβαστική. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 57-58 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 63 υπέρ Πάμε στην 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 71-72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 73 υπέρ το ΕΚ πώς ψηφίζει Ποιος είναι κατά. Εγκρίνεται. 74 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχεται. Παρακαλώ συνάδελφοι να συμμετάσχετε όλοι στην ψηφοφορία γιατί αλλιώς ε, επιμηκύνουμε όλη τη διαδικασία και κάνουμε αυτή την ηλεκτρονική ψηφοφορία που μας ε, κάνει να καθυστερούμε. Πέρα της ψηφοφορίας. 31 υπέρ, 33 κατά, απορρίπτεται. Ποια ήταν αυτή η 74. Ωραία, πάμε στην 75. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται οπότε τώρα 78-79-80 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 81 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 82 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 83 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 84 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται απορρίπτεται ελέγχουμε Πέρας της ψηφοφορίας 25 υπέρ, 36 κατά απορρίπτεται πολύ αντέχει σήμερα ο κύριος Μπουτικόφερ. Απίστευτο. Σόλτ, 86 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 87 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 88 υπέρ. Κατά. Αποχές να ελέγξουμε. Όχι, μάλλον απορρίπτηκε, απορρίφθηκε. 89 υπέρ. Κατά απορρίπτεται 90 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 92 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 95, 94 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 95 υπέρ. Κατά. Αποχές ελέγχουμε. Νομίζω ότι εγκρίνεται βέβαια. Abstimmung ist geschlossen. Πέρα τη ψηφοφορία. 42 υπέρ, 25 κατά εγκρίνεται, 96 υπέρ, κατά. Παρακαλώ άλλη μια φορά, την 96 υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 97 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 98 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 100, 101, 102, 103 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε αλλά αν και νομίζω ότι εγκρίνεται εγκρίνεται με 38 υπέρ και 29 κατά. Πάμε στην 106 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 107 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 108 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 109 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 110 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 111 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 112 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 113 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 114 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 115 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 116 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 117 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 118 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 119 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 120 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 121 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 122 και 123 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 124 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 125 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 126 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 127 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 128 129 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 130 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 131 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 132 και 33 υπέρ, κατά, αποχές, ελέγχουμε. Πέρα της ψηφοφορίας. 32 υπέρ, 34 κατά, απορρίπτεται. 134 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 135 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 136 υπέρ, συγγνώμη, 137 ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 138 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 139 υπέρ κατά αποχές απο, εγκρίνεται 140 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 141-142 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 143 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 145 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 146 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 147 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 150 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 152 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 154 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 155 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και πάμε τώρα στις ε, τροπολογίες 2, 3, 4. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 11 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται.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 αποχές απορρίπτεται. 27, 28 και 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 30 και 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 33, 34, 35. Πολύ πάλι ενδιαφέρουσα η συμμαχία. Ο συνδυασμός μάλλον. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ο κύριος Λάινεν <coughs> Um ganz korrekt zu sein, sollten wir den 194 noch για να είμαστε σωστοί πρέπει να ψηφίσουμε και την 194 γιατί 98 και 99 ε, δεν ε, βγήκαν επειδή είχαμε λίγο δύο παραπάνω στο ΕΛΚ. Για να είμαστε σωστοί λοιπόν πρέπει να ψηφίσουμε και αυτοί. Είμαστε στο σημείο που είχαμε πει ότι υπήρχε διόρθωση γιατί είχαμε διαφορά έξι ε, ψήφους, μετά τελικά ήταν τέσσερις, οπότε αυτό αποφασίστηκε. Για την 194 όχι. Το προσέξαμε, δεν ήταν δύο παραπάνω, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα, απλώς το είπατε εσείς από το βήμα. Το είπα σε μία περίπτωση που ήταν 36 με 32. Ούτως ή άλλως υπήρχε πλειοψηφία από την άλλη πλευρά και δεν υπήρχε νόημα. Εντάξει, δεν ήταν τόσο ξεκάθαρο, τώρα μου το ξεκαθαρίσατε. Ευχαριστώ. Πάμε λοιπόν στο τέλος. Περνάμε λοιπόν στην ε, τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Παρακαλώ να ψηφίσουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Λοιπόν, με 52 υπέρ, 5 κατά και 9 αποχές ε, πέρασε, υπερψηφίστηκε η έκθεση Συγχαρητήρια λοιπόν στον εισηγητή και στους ε, σκιαδησηγητές ε, και πιστεύω ότι αυτή η αναβολή που είχαμε ζητήσει είχε νόημα γιατί μπορέσαμε να τα ξαναπούμε. Βέβαια η ώρα εντωμεταξύ έχει πάει 10 και πρέπει να φύγουμε από την αίθουσα που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση για την Βενεζουέλα. Θα τα πούμε την επόμενη φορά, ε, το αργότερο 7 ε, Δεκεμβρίου μετά τις εκλογές.